στο θέμα αυτό. Σημαντικά μέτρα λοιπόν έχουμε πλέον ε, δώσει την κατεύθυνση για να έχουμε ένα πιο ασφαλή εφοδιασμό στο μέλλον. Αλλά αυτό είναι ένα βήμα μόνο προς την κατεύθυνση της Ενεργειακής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που συμμετείχαν στη συζήτηση, η οποία αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία επί της εκθέσεως Μπούζεκ θα πραγματοποιηθεί